Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Συνεχίζουμε με τη σημερινή μας συνεδρίαση και αυτή τη φορά έχουμε προσκεκλημένο τον κύριο Τεκρέμ, ο οποίος είναι Υπουργός Άμυνας του Βελγίου έρχεται συχνά στην Επιτροπή μας και ο κύριος Ποπόφσκι είναι μαζί για την εξωτερική δράση και αυτός έρχεται συχνά στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε λοιπόν για να μας μιλήσετε για τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων υπό τη σύνθεση των Υπουργών Άμυνας που έλαβε χώρα τη Δευτέρα που μας πέρασε στις Βρυξέλλες. Είχαμε και τον Επίτροπο Φίλε και τον κ. Πινιόν που είναι ο Ιωνικό Γραμματέα τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση, όπου ακούσαμε για την εξωτερική δράση. Σήμερα έχουμε την άμυνα. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα εδώ που έχει να κάνει με τις διάφορες ε, δράσεις μας, τις αποστολές μας. Όπως επίσης είναι και το θέμα των, ε, της ανάπτυξης δυνατοτήτων και αυτό είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πολύ. Υπάρχουν και διάφορες πρωτοβουλίες, Οι ειδικοί και άλλες. Πολλές πρωτοβουλίες ακούγονται τελευταία με το περίφημο pooling and sharing, που είναι όρος ε, πολύ της μόδας, που είναι η συγκέντρωση και η αποκοινού χρήση δυνατοτήτων. Να λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αυτά είναι τα δύο μεγάλα κομμάτια των θεμάτων που θα θέλαμε να μας αναπτύξετε. Θέλω να προσθέσω επίσης εδώ και κάτι ακόμα γιατί είναι ένα θέμα που θα μας ενδιαφέρει και στο μέλλον. Πήγαμε στην Ουγκάντα, μια, υπο, μια αντιπροσωπεία της υποπιτροπής μας πήγε εκεί και καταλήξαμε σε θετικά συμπεράσματα, δηλαδή εντυπώσεις μας ήταν θετικές και όσον αφορά τις τεχνικές δυνατότητες της αποστολής μας εκεί, αλλά και όσον αφορά ε, τους πολιτικούς λόγους, το πολιτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για την αποστολή εκεί. Ήταν θετικέ οι εντυπώσει μα δηλαδή από αυτήν την επίσκεψη στην εκεί αποστολή μα. Έχετε το λόγο χωρί άλλη καθυστέρηση, κύριε Υπουργέ. Αγαπητοί συνάδελφοι της Επιτροπής, ε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολύ χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία να βρεθώ εδώ σήμερα μαζί σας για να σας μιλήσω για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπό τη σύνθεση των Υπουργών Άμυνας που έλαβε χώρα τη Δευτέρα. Η Άστον δεν είναι εδώ σήμερα και μου ζήτησε να την αντικαταστήσω, οπότε ευχαρίστω θα την αντικαταστήσω. Πριν μπω στην ουσία της συνάντηση, θέλω να σα πω ότι είναι τρίτη φορά που το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ε, συνεδρίαση υπό τη σύνθεση των Υπουργών Άμυνας και οι Υπουργοί Άμυνας επίσημα ε, κατέληξαν σε συμπεράσματα και διοθέτησαν. Άρα πια η σύνθεση αυτή αποτελεί ανακεκτημένο. Οι επίσημες αυτές συνεδριάσεις των Υπουργών Άμυνα ε, αποδεικνύουν ότι η κοινή πολιτική ασφάλεια και Άμυνα πια έχει εδρεωθεί και δείχνει επίση και την επιλογή τη ΥΠΑ του εκπροσώπου για τη σημασία που έχει η σύνθεση αυτή για γενικότερα την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα λοιπόν τώρα από αυτό να αναφερθώ στο Συμβούλιο αυτό καθευτό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την εφαρμογή της εθήκης της Λισαβόνας που είναι στο κέντρο των προσπαθειών μας και όσον αφορά την ε, ΚΕΠΑ και όσον αφορά την ολοκλήρωση και όσον αφορά τις αποστολές μας που αποτελούν μέρος του, της εργαλειοθήκης όπως τη λέμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δύο λόγια, πιστεύω ότι πρέπει να περάσουμε τώρα στην λειτουργική πραγματικότητα. Έπειτα, πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, βλέπουμε αλλαγές στις γείτονες χώρες, με αποτελέσματα τα οποία είναι ακόμα ασαφή. Έτσι λοιπόν, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κυβερνήσεις ε, προσπαθούν ε, επιπλέον να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Και μέσα εδώ μπαίνει και ο προπολογισμό άμυνας των διαφόρων χωρών. Θα περιοριστώ στην συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας και γι' αυτό θα σας αναφέρω κάποια στοιχεία όσον αφορά τις, ε, την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων μας και τις αποστολές μας, αλλά και θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής και άμυνας και τέλος θα κοιτάξουμε λίγο τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Οι αποστολές της CSDP, της ΚΕΠΑ δηλαδή, θέλουν να περάσουν στην πράξη επιτόπου. Οι συνάδελφοι και εγώ έχουμε συζητήσει τις διάφορες τέτοιες αποστολές Πολλέ φορέ και την παρουσία των απληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Και ένα από του λόγου που το κάναμε αυτό είναι γιατί πολύ συχνά κοιτάμε τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ από θεσμική οπτική γωνία. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι λειτουργούμε δίπλα ένα στον άλλον σε πάρα πολλού χώρου και στη Σομαλία και στο Αφγανιστάν και στα Βαλκάνια. Και αυτό το, αυτή η σχέση είναι κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Είναι ζωτική σημασία. Η καταπολέμηση της πειρατείας, για παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, εξακολουθεί να είναι πηγή ανησυχία. Η Αταλάντα, η αποστολή μας αυτή είναι επιτυχής, αλλά ο τρόπος που λειτουργούν οι πειρατές αλλάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δράσει για να κάνει κάτι για αυτό το θέμα. Με αποτέλεσμα να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει έγκριση αλλαγών όσον αφορά τη δράση μας εκεί. Πολλές χώρες μέλη επίσης ζητούν μια πιο έντονη δράση. Αλλά υπάρχουν νομικά ζητήματα τα οποία παραμένουν στην ημερήσια διαταξή μας, ιδιαίτερα η μεταφορά των υπόπτων πειρατών. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να υπογράψει μια συμφωνία με την Σομαλία. Θα πρέπει επίσης να βρούμε μια πιο βιώσιμη λύση. Η το εκπρόσωπος θέλει συμφωνίες με τις διαφερόμενες χώρες ώστε να μπορέσουμε με τη σειρά μας να ενισχύσουμε τις προσπάθειες που κάνουν για την καταπολέμηση της πειρατείας οι χώρες αυτές στην περιοχή. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η αποστολή Αταλάντη όσον αφορά τους Σομαλούς στρατιώτες στην Ουκάντα είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αντιπροσωπεία της Υποπιτροπής Άμυνας και ασφάλειας που ότι πήγε στην Ουγγάντα, επισκέφθηκε την αποστολή μας αυτή και στον Πιάνκα όπου βρεθήκατε αλλά και στην Καπάλα. Πολύ θα ήθελα να ακούσω τις εντυπώσεις σας. Είναι πολύ σημαντικές για μας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν μέσα στους επόμενους μήνες αν θα παραταθεί ή όχι η αποστολή αυτή. Υπάρχει μια τάση να επαναπροσανατολιστεί η δουλειά της αποστολής στη δημιουργία μιας, ε, ε, ε, μιας βοήθειας προς τις αρχές. Για τους υπουργού Άμυνα ήταν η ευκαιρία να δώσουν ήδη κάποιους προσανατολισμούς στο Συμβούλιο αυτό που πέρασε. Πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε από κοντά τι γίνεται με τους στρατιώτες που εκπαιδεύουμε. Και αυτό ισχύει και για την Αταλάντη και για το UTM. Πρέπει να συζητήσουμε για το μέλλον των αποστολών μας στα πλαίσια μιας περιφερειακής προσέγγισης ευρύτερης, στο κέρας της Αφρικής για παράδειγμα, για να έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση η οποία συμπεριλαμβάνει όλα τα μέσα που διαθέτει η Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τελευταία, η ίδια μάλλον παρατήρηση ισχύει και για την αποστολή μας Αλτέα στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την παρουσία των δυνάμεών μας στη χώρα αυτή. Η κατάσταση είναι ανησυχητική ακόμα και αν δεν πρόκειται για θέματα ασφάλειας αυτά κάθε αυτά. Οπότε η ύπατος εκπρόσωπο ζήτησε από τους Υπουργού να συνεχίσουν να στηρίζουν την αποστολή αυτή. Η παρουσία τώρα εκπροσώπου του ΝΑΤΟ ήταν κάτι πολύ χρήσιμο στη συζήτηση που κάναμε για την ΕΟΦΟΡ στην Λιβύη. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε έναν ε, επικεφαλής της αποστολής και ολοκλήρωσε και το σχεδιασμό για μια αποστολή ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να δράσουμε μετά από το αίτημα των Ηνωμένων Εθνών για να συντονίσουμε τις ανθρωπιστικές υποθέσεις εκεί. Η το εκπρόσωπος μετά την επίσκεψή της στη Βεγάζη επέμεινε προς τους ε, υπουργούς ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε γρήγορα στις προκλήσεις που τίθενται εκεί. Είναι σαφές, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η ΕΦΟΡ, εφόσον ξεκινάει συνεργασία με το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ, μην ξεχνάμε ότι ελέγχει και τον ενέργειο και το θαλάσσιο χώρο, οπότε χρειάζεται μια τέτοια συνεργασία. Απ' την άλλη, ούτε το ΝΑΤΟ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ενδείξει ότι θα συζητηθεί συντονισμός των ανθρωπιστικών υποθέσεων άμενα, άμεσα. Εκ παραλλήλου γίνεται βέβαια σχεδιασμός και από τον ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό χρησιμοποίησαμε αυτή την ευκαιρία για να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερο τους δύο οργανισμούς μεταξύ τους. Και ε, μιλήσαμε για ε, συνάντηση των δύο αυτών πλευρών προκειμένου να συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα το θέμα της Λιβύης. Έρχομαι τώρα στο σχεδιασμό. Για να στηρίξουμε τη Λιβύη πιο μακροπρόθεσμα στην περιοχή, προβλέπουμε μια αναθεώρηση του τομέα της ασφάλειας. Έχει ξεκινήσει αυτό υπό την ηγεσία της ΥΠΑ του εκπροσώπου. Ένα άλλο θέμα, Πρόεδρε, το οποίο επίστησε την προσοχή μας, είναι το θέμα των στρατιωτικών δυνατοτήτων, κάτι που σε καλά γαλλικά λέει ο μιλητής, θα λέγαμε pooling and sharing. Πώς δηλαδή θα βάζουμε μαζί τις δυνάμεις μας και από κοινού θα τις χρησιμοποιούμε. Για πρώτη φορά αναλύσαμε μαζί τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, τις δυνατότητες άμυνας που έχουμε. Και έτσι καταλήξαμε σε μια κοινή πρωτοβουλία από τη Γερμανία και την Σουηδία. Και οι υπουργοί συμφώνησαν για ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα το Δεκέμβριο του 2010 όπως το υπογραμμίζει και η προσωρινή έκθεση της ΥΠΑ του εκπροσώπου για την πολιτική ασφάλειας και Άμυνας που παρουσιάστηκε στους υπουργού Άμυνας και λέει ότι εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να παραμείνει ενεργό στοιχείο στον κόσμο θα πρέπει να έχει ε, σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες. Όμω, στα πλαίσια που βρισκόμαστε σήμερα, στο οικονομικό πλαίσιο δηλαδή, υπάρχει κίνδυνο να μειωθούν οι στρατιωτικέ αυτέ δυνατότητε. Έτσι λοιπόν η αμοιβαιότητα ή ο διαμερισμός των δυνατοτήτων αποτελούν μέρος της λύσης. Η συνάντησή μας αυτή επιβεβαίωσε ότι υπάρχει πολιτική βούληση προκειμένου να βρούμε νέο ε, δυναμισμό για τη διαδικασία αυτή. Έχει ήδη γίνει πολλή δουλειά. Όλες οι χώρες μέλη έχουν συνεισφέρει με ιδέες και έχουμε πάνω από 300 δυνατότητες, προτάσεις δηλαδή επιτάπητος. Πολύ καλό αποτέλεσμα αυτό, αξιοσημείωτο. Τώρα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε ώστε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και σε πολιτικό επίπεδο βέβαια. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες αυτές είναι ρόλος ε, ε, καταλυτικός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θέλουν περισσότερη διαφάνεια για να εντοπίζονται οι δυνατότητες που υπάρχουν για σχέδια στο μέλλον, να εντοπίζουν ποια είναι τα στοιχεία της επιτυχίας και είπα εκπρόσωπος φυσικά και είναι έτοιμη να συνεχίσει να βοηθάει και να ενισχύει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον το επιθυμούν τα κράτη-μέλη. Συγχρόνως όμως είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν για τη διαδικασία αυτή, να την νιώσουν δικιά τους, να παίρνουν αποφάσεις, γιατί τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που έχουν τις δυνατότητες τελικά. Νομίζω ότι συμφωνήσαμε όλοι για τον κεντρικό ρόλο που έχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Αυτή η αμοιβαιότητα και η συγκέντρωση και από κοινού χρήση των ε, πόρων είναι το βασικό στοιχείο. Τώρα, επιπλέον, 17 Υπουργοί υπέγραψαν συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Στόλο Στρατηγικών Μεταφορών. Η ύπατος εκπρόσωπος υπενθύμησε, και αυτό τώρα το λέω στα πλαίσια του Benelux, είπε ότι θα συνεχίσει να φροντίζει να επεκταθούν τα ήδη υπάρχοντα σχέδια ή να προσθεθούν και νέα. Και μετά από ερωτήσει των συναδέλφων θα δείτε στο παράρτημα ότι γίνεται μία για μια έκτακτη συνάντηση όπου οι Υπουργοί μπορεί να ανακοινώσουν νέε αποστολέ, νέε δεσμεύσει που αναλαμβάνουν. Αυτό μέχρι τα τέλη της χρονιάς ή το 2012 ανάλογα με την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί. Τέλος, η ότι εκπρόσωπος υπενθύμησε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τις προσπάθειες που κάνει το ΝΑΤΟ. Χρειάζεται άμεση συνεργασία. Και πολλοί υπουργοί τη στήριξαν σε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τους τελευταίους μήνες είδαμε πολλές αλλαγές στα κράτη-μέλη. Και... Στον τομέα που μας απασχολεί σκέφτομαι παραδείγματο χάρη ε, την ε, επιστολή και την ε, στάση των Βρετανών συναδέλφων που αποδεικνύουν περισσότερο pooling and sharing για να υπάρξει μία θετική πρόοδο. Στα πρέσια αυτά λοιπόν το θέμα της, ε, ε, των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, έχει έχει ε, τονιστεί ιδίως ε, στις συζητήσεις με πολλούς ε, υπουργού και στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφαλείας πρέπει να προγραμματίσουμε πόσο θα διεξάγουμε τις αποστολές, πώς θα τις προγραμματίζουμε με στόχο την αποτελεσματικότητα και το σημείο κινήσεως είναι να αξιολογήσουμε τις ανάγκες μας, τι χρειαζόμαστε και τι έχουμε σε σχέση με τις ανάγκες ε, οι οποίες διαμορφώνονται. Ε, και το πρόβλημα ε, χρειάζεται πιο λεπτομερή εξέταση βάσει των μαθημάτων που έχουμε αποκομίσει από προηγούμενες αποστολές. Θα ήθελα στο τέλος να αναφερθώ και στο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού διότι ε, διευθύνεται από την κάθε Άστον ε, και πλέον της αρχής του pooling and sharing και συζητάμε ένα θέμα το οποίο επίσης χρήζει προσοχής δηλαδή την ε, επίπτωση των πολλαπλών πολιτικών αμήνης στην Ευρώπη και αναφέρομαι στον ενιαίο ο ουρανό της Ευρώπης που θα επηρεάσει τους στρατιωτικούς και ε, το γραφείο μας ε, προσπαθεί να βοηθήσει σε μια ενιαία διατύπωση αυτού του στόχου και όσον αφορά τις ε, επόμενες, τους επόμενους μήνες ελπίζω ότι το pooling and sharing θα παραμείνει στο επίκεντρο του έργου των Υπουργών. Δεν θέλω να υπερβάλλω αλλά ε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και ε, όλοι οι Υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως συμφωνούν ότι πρέπει να διατηρηθεί ε, μη ένα υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας για να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Πολλά θέματα θα συζητηθούν από τους υπουργούς όπως ε, το θέμα των συνεργειών μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών συνεργασιών όχι μόνο με το ΝΑΤΟ αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με την, Αμερικα... με την Αφρικανική Ένωση και ε, θα σας ε, παρουσιάζουμε τις ε, εκθέσεις εκτενώς σε ένα σύνολο το οποίο θα προωθηθεί τον Ιούλιο και θα παρουσιαστεί κατά τρόπον ώστε να προωθήσουμε τη δράση μας. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτές, επαναλαμβάνω ότι χαίρομαι ιδιαίτερος που μπόρεσα να σας ενημερώσω για την έκβαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων εν ονόματι της είπα της εκπροσώπου και ε, προσλέπω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την πολύ πλήρη αυτή εικόνα που μας παρουσιάσατε. Ε, Βλέπετε εδώ κινούμε σαν στρατιωτικός με την πειθαρχία που επιβάλλεται. Είστε πολύ αποτελεσματικός λέει ο πρόεδρος. Υπάρχουν διάφορες ενδιαφέρουσες βάσει, ιδίως κατόπιν της αποστολής στη Βενγάζη και θα ήθελα να σας πω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετήσαμε την ετήσια έκθεση για την ε, κοινή πολιτική που ε, φέτος συνέταξε ο Ρομπέρτο Γκαλτιέρη ε, που στήριξε τον προηγούμενο μήνα, μάλλον αυτό το μήνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Άρα όλοι είμαστε ε, πεπισμένοι για την ε, αναγκαιότητα αυτής ε, της κοινή πολιτικής η οποία λειτουργεί καλά ακόμη και αν προς το παρόν έχει περιορισμένο ρόλο και είναι μία φιλοδοξία την οποία πρέπει να υλοποιήσετε. Στηρίζουμε λοιπόν πάρα πολύ την πολιτική αυτή και πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές ε, ε, δεν βλέπουμε να αντικατοπτρίζεται στο πολιτικό επίπεδο από τα κράτη και από την ύπατη εκπρόσωπο και ε, γι' αυτό πολλές φορές αισθανόμαστε κάπως απογοητευμένη και η απογοήτευση αυτή ιδιαιτέρως εξεφράσει στα πλαίσια της Λιβύης διότι το ψήφισμα του Μαρτίου του Κοινοβουλίου προέβλεπε ορισμένες διατάξεις οι οποίες δεν ήταν πολύ ε, ε, ε, φιλόδοξες αλλά μπορούσαν να υλοποιηθούν στο θαλάσσιο τομέα και στο τομέα του εμπαργο και απογοητευθήκαμε διότι είδαμε ότι δεν υλοποιήθηκαν τα μέτρα αυτά και τελικά βασιστήκαμε στο ΝΑΤΟ για τις επιχειρήσεις αυτές ενώ εμείς ζητούσαμε πέραν των αεροπορικών υπεθέσεων να υπάρξει και μία παρακολούθηση στα θαλάσσια. Οπότε θα έπρεπε τώρα να αποκομίσουμε τα συμπεράσματα, να κοιτάξουμε την υπόθεση αυτή και να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα συμπεράσματα σχετικά με τη Λιβύη και την κοινή πολιτική ασφαλείας και αμήνης. Τέλος, ε, ε, σχετικά με τις δράσεις που αναφέρατε και θεωρήσαμε ότι ήταν επιτυχής το πρώτο θετικό σημείο ήταν ότι η τελευταία αυτή αποστολή οικονομικά ήταν περιορισμένη και μας ε, προσέφερε ωφέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την κρίση στη Σομαλία, στο κέρας της Αφρικής και ε, πρέπει να την αξιολογήσουμε θετικά. Επίσης ε, διαπιστώσαμε και ορισμένες ελλείψεις και αυτό που μας ε, εκπλήσει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει ένα βασικό μέρος την εκπαίδευση των στρατιωτών επί εβδομάδες στην Ουγγάντα χωρίς να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει προς τα πίσω πώς επιλέγονται οι νεοσύλλεκτοι και στη συνέχεια πώς χρησιμοποιούνται. Πιστεύουμε λοιπόν ότι εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει την εκπαίδευση θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τους ανιώντες και κατιώντες, τις ανιούσες και κατιούσες διαδικασίες δηλαδή καταρχήν εφόσον είχαμε 900 νεοσύλλεκτους από την Σομαλία είδαμε ότι εξ αυτών 100 ε, επιστράφηκαν στη Σομαλία διότι οι γιατροί δεν τους θεώρησαν ε, ως ε, καταλήλους. Ε, ορίστε λοιπόν ορισμένα πράγματα τα οποία σημειώσαμε χωρίς βέβαια να αμφισβητούμε την πολιτική σημασία αυτής της αποστολής και τον επαγγελματισμό των επιτόπου εμπλεκομένων. Αυτά είχα να σας πω και ε, θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις σε ερωτήσεις αυτές. Ξεκινάει όμως η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να μιλήσω για τη Λιβύα. Λιβύη. Συμμετείχα σε ε, αυτή την αποστολή ε, στη Βενγάζη από τις 17 στις 20 Μαΐου και μπόρεσα και εγώ να μεταβώ στις, ε, στην πρώτη γραμμή νοτίως της Βενγάζης σε μερικά χιλιόμετρα δυτικά όπου υπάρχουν 3.000 στρατιώτες του Καντάφη ε, τους οποίοι, οποίοι κοιτάζονται με τους 1.400 ε, στρατιώτες των ε, επαναστατών. Υπάρχει ένας ε, λόφος ε, που ακολουθεί την ε, παραλία και εκεί διεξάγονται οι αναμετρήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κόσμος αυτός είναι πολύ κακά οπλισμένος, υπάρχουν στην πρώτη γραμμή άτομα που δεν έχουν καν ε, μπότες που φορούν σάνδαλα και ε, μπλουζάκια, t-shirt. Δεν έχουν στολές. Και οι περισσότεροι είναι νέοι. Νέοι που ποτέ δεν έχουν εκπαιδευτεί στρατιωτικά που ήταν ε, γιατροί, μηχανικοί, έμποροι, δάσκαλοι και ούτω καθεξής. Μου είπα, μας είπαν λοιπόν ότι εκτιμούν ιδιαίτερο τη δράση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, του ΝΑΤΟ και είναι καταφανής ε, η η ευγνωμοσύνη αυτή με πόστερς πάνω στα αυτοκίνητα. Θέλω όμως να επισημάνω ότι θα μπορούσε να υπάρξει μία καλύτερη διασύνδεση με το ΝΑΤΟ διότι υπάρχουν ορισμένοι Λίβοι οι οποίοι έχουν αποσχεθεί από το καθεστώς και ε, ηγούνται των επιχειρήσεων χωρίς να έχουν όμως απάντηση σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχουν στον ΝΑΤΟ σχετικά με τους χώρους όπου θα μπορούσαν να, επιτεθούν ή να πλήξουν. Είδα λοιπόν πώς εργάζονται. Ε, εργάζονται βάσει των πληροφοριών που δίνει ο λαός, λέγοντας είδαμε αυτό, εκείνο το άλλο. Έχουμε όμως ένα ε, κέντρο με δορυφόρους που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο και που έχει διατεθεί σε άλλες επιχειρήσεις. Οπότε γιατί όχι, γιατί να μην χρησιμοποιηθεί και εδώ. Και βεβαίως νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε γιατί ο, ο λαός της Λιβύης είναι οπλισμένος και μάχεται. Σε αυτά συμφωνώ με τον Πρόεδρο. Είμαστε απογοητευμένοι ότι η αποστολή που είχαμε ζητήσει με το ψήφισμα της 10ης ε, Μαρτίου δεν έχει γίνει. Ε, μας είχαν πει ότι θα γινόταν ε, αλλά ήταν πρωταπληλιάτικο αστείο, δεν υλοποιήθηκε. Το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει να μπορέσει να εφαρμοστεί το εμπάργο των οπλισμών που είναι πολύ σημαντικό και ιδίω διότι έπρεπε να επιτηρούνται και τα τεράστια σύνορα της Λιβύης ιδίως νοτίως προς τον νότο διότι από εκεί θα μπορέσουν να διεισδύσουν οι τρομοκράτες και γνωρίζουμε ότι γείτονες σαν την Αλγερία και το Τσάντ και, το, και ο Νίγηρας παίζουν κάποιο πολύ αμφιλεγόμενο ρόλο. Δεν ε, μιλάμε λοιπόν μόνο για την ε, Λιβύη αλλά και για εμάς. Και έπρεπε αυτή η ε, αποστολή να γίνει για να εφαρμόσουμε αυτό που μας ζήτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας, να προστατεύσουμε ε, τους ε, Λίβιους. Αλλά ε, από την άλλη πλευρά ε, υπάρχει μια σημαντική εμπλοκή ανθρωπιστική μέσω του προγράμματος ΕΚΟ όλα, ε, όλες οι ανθρωπιστικές προσπάθειες έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επιγόντως θα έπρεπε συγχρόνως να υπάρξει και μία προστασία των ε, περιοχών που βρίσκονται στις ε, δυτικές παρυφές ε, της, της όπου υπάρχουν βερβέροι και κοινότητες όπου παραπονούνται ότι δεν έχουν ούτε νερό ούτε ιατρική βοήθεια και άρα νομίζω ότι αυτή η αποστολή είναι τώρα προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να την αναπτύξουμε με τη βοήθεια των αρχών της Τινησίας. Και αυτός, αυτή η αποστολή δεν έχει μόνο στόχο να προστατεύσει τους πολίτες όπως μας το ζητά το Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά αν βλέπατε το CNN σήμερα το πρωί, ε, ε, βλέπαμε τα παιδιά τα οποία τα βάζουν μέσα σε σπηλιές για να ζήσουν υπό φοβερές και απαράδεκτες συνθήκες υπάρχει και ε, μία πολιτική, ένα θέμα πολιτικής ισχύω. Ε, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση των δυνατοτήτων ε, της κυβερνήσεως του Καντάφη αλλά υποφέρει ο πληθυσμός της Τρυπόλεως και λυπούμε πάρα πολύ διότι τα κράτη-μέλη κρύβονται πίσω από το θέμα αυτό και δεν αναπτύσσεται αυτή η αποστολή ε, της CSDP διότι αντιλαμβάνομαι ότι αυτοί που είναι επιτόπου δεν γνωρίζουν ακριβώς τι χρειάζεται και από την άλλη πλευρά υπάρχουσε, τα υπάρχοντα ψηφίσματα του ΟΗΕ μας δείχνουν τον δρόμο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει πιο σαφής αποστολή για την USDP από αυτήν. Και τέλος, ε, και πιστεύω ότι αυτό συμφωνεί με αυτά που είπατε, ε, χρειάζεται να καταρτιστεί μία νέα αποστολή για να μπορέσουν όλοι αυτοί οι νέοι οι οποίοι βρίσκονται ε, τώρα στα checkpoints πίσω στο χώρο τους. Ευχαριστώ Άννα. Έχουμε μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, οπότε σας παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι για να έχουμε και απαντήσεις. Ο κύριος Κόβατσεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή σας παρουσία εδώ. Θα ήθελα να θυμηθούμε κάτι πονίδιστο βέβαια, αυτό που συνέβη στη δεκαετία του 50 με την απόρριψη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άμυνας και βλέπουμε ότι πλέον ε, η συγκέντρωση και ανταλλαγή των πόρων μας, το pooling and share, ε, βρίσκεται πλέον στην προτεραιότητα των ε, αναγκών μας. Ε, βέβαια, εντάξει, αυτά είναι παρελθόν, δεν έχει και τόση σημασία πια που απερίφθη τη δεκαετία του 50, απλώς ως υπενθύμηση το είπα. Κατά την άποψή σας, κύριε Υπουργέ, πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει η διαδικασία και να έχουμε κοινέ δυνατότητες. Αναφέρατε, αν άκουσα καλά, 300 δυνατότητες ε, πόρων αυτού του pooling και sharing. Έχουμε διάφορες δομές τώρα, υπάρχουν ε, το Eurocorp, υπάρχουν κάποιες ιδέες για να υπάρχει κάποιος εξοπλισμός ε, σε κατάσταση αναμονής για χρήση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη διάθεση κάποιων κρατών μελών. Θεωρείτε όμως ότι διμερείς συμφωνίες όπως αυτή που έκανε η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ή μεταξύ Γερμανίας και Σουηδίας είναι η κατάλληλη απάντηση ή χρειαζόμαστε κάτι πιο υπερεθνικό υπό τη σκέπη και της ε, κοινή ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και αυτής της δομής του pooling and sharing. Όσον αφορά τώρα αυτά που ανέφερε και η κυρία Γκόμες για τη Λιβύη, Πολλοί λένε ότι η ζώνη απαγόρευση πτήσεων δεν είναι λύση, είναι απλώς ένα πρώτο βήμα, πρέπει να δράσουμε και επιτόπου αν θέλει κάποιος να έχει επιτυχές αποτέλεσμα στη Λιβύη. Θεωρείτε ότι η κατάλληλη επιλογή είναι να εξοπλίσουμε τους επαναστάτες ε, με όπλα, επαρκεί αυτό. Ε, υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι έχουμε πικρά πείρα με τους Μιτζαχεντίν στο Αφγανιστάν, τους εξοπλίσαμε και μετά γίνανε λιμπάν και ε, πολεμούν εμάς. Ελπίζω να μην συμβεί και εδώ το ίδιο. Ελπίζω οι υπηρεσίες πληροφοριών μας να γνωρίζουν ε, ε, τι ακριβώς κάνουν οι επαναστάτες στη Βεγγάζη και αυτό το προσωρινό συμβούλιο. Ε, θεωρείτε ότι χρειαζόμαστε μια αποστολή επιτόπου εκεί. Ο κύριος Κάμπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο πράγματα. Καταρχάς, την περασμένη εβδομάδα ήμουν στην Ταϊβάν, ε, μίλησα με τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και τον Επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας. Να πω εξ αρχής ότι είμαι φίλος της Ταϊβάν και ε, υποστηρίζω την κυβέρνηση της Ταϊβάν. Υπάρχουν όμως και εκεί θέματα ασφάλειας και άμυνας, ε, υπάρχουν υποβρύχια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και δεν μπορούν να βρουν κάποιον να τους βοηθήσει να έχουν πιο σύγχρονα υποβρύχια για, το, ε, για την άμυνά τους. Ένα εξ αυτών χρονολογείται από το 1943. Επίσης ε, θέλουν περισσότερα και πιο σύγχρονα F-16. Το θέτω αυτό γιατί μιλάμε για ξένες αποστολές που σχετίζονται με την άμυνα και ίσως μπορεί να μας ενδιαφέρει. Τώρα, για να περάσω στα όσα έλεγε ο Υπουργό. Μιλήσατε για φιλοδοξία και είπατε ότι πρέπει να έχουμε υψηλέ προσδοκίε. Το επίπεδο φιλοδοξιών όμως ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας είναι να έχουμε έναν ε, νέο ευρωπαϊκό στρατό. Και επίσης να πω το εξή. η Βαρόνια Άστον ήταν κατά της ζώνης απαγόρευσης πτήσης. Εγώ την αποκαλώ η κόκκινη Βαρόνη γιατί προσπάθησε να, το, να την κλείσει. Ε, είστε εσείς υπέρ αυτής της διόνυσης απαγόρευσης πτήσεων που υποστήριξε ο Ντέιβιτ Κάμερον με τόσο σθένος. Ευχαριστώ και συγγνώμη αν καθυστέρησα αν ρωτήσω πράγματα τα οποία έθιξε ήδη ο κύριος Ντεκρέμ. τότε θα ρωτήσω τους συναδέρφους για να μου πούν τι υπόθηκε σχετικά. Το ένα είναι η Αταλάντα. Θέλω να αναφερθώ στην αποστολή Αταλάντα η οποία είναι μια δυνατή, μια καλή αποστολή. Στην πράξη, τι έχει γίνει, υπάρχει καμιά αλλαγή στην, ε, στους όρους. Βλέπετε, εμείς έχουμε κάποιους ε, δισταγμούς για το κατά πόσο είναι η σωστή αυτή λύση να πιάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους πειρατές και να τους πηγαίνει στο δικαστήριο. Ε, μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ακόμα καλύτερο γιατί τελικά τι σημαίνει αυτό ότι έχει αποτύχει η μέχρι τώρα αποστολή μας. Γιατί εδώ έχουμε τον πόλεμο κατά της πειρατείας. Και κάτι ακόμα για την U4 στην Λιβύη. Το σχέδιο αποστολής έχει εγκριθεί ήδη. Και τι περιλαμβάνει, τι μπορείτε να μας πείτε για το ποιες χώρες είναι διατεθειμένες να προσφέρουν ποιες δυνατότητες και τι προσωπικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Γουαλτιέρη. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα είπε ο πρόεδρος Νταρζάν για την έκθεση που εγκρίναμε και τη σημασία της, ε, η οποία είναι και πολιτικής ε, φύσεως, διότι έτυχε και αθρώας υποστήριξης, ε, που σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει αναλάβει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δέσμευση να υποστηρίξει την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμενας και θέλει να είναι συνομιλητής και με το Συμβούλιο και με τους Υπουργούς Άμυνας και θεωρούμε ότι πρέπει και να υπάρχει ένας υπουργό άμυνας που να έχει αυξημένο ρόλο. Αναφερθήκατε σε αυτό το συμβούλιο, το οποίο μάλλον ήταν αρκετά πιεσμένο χρονικά. Για το pooling και sharing, χαιρόμαστε που αυτή η έννοια που ξεκίνησε πριν από κάποιο διάστημα είναι πλέον κεκτημένο, αν μου επιτρέπετε την έκφραση δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αν μου επιτρέπετε, αν τα περαιτέρω βήματα που γίνονται είναι βήματα τα οποία θα μας οδηγήσουν σε μια επιχειρησιακή φάση ή αν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και δεν μπορούμε να περάσουμε πιο συγκεκριμένα στην επιχειρησιακή φάση. Θα ήθελα λοιπόν και τη δική σας την εκτίμηση επ' αυτού και κάποια στοιχεία για τις πιο μεγάλες χώρες οι οποίες θεωρώ ότι αποτελούν ικανή και αναγκαία συνθήκη για να έχουμε μία πιο σωστή τοποθέτηση και εφαρμογή του pooling and sharing. Κάποια στοιχεία επιπλέον λοιπόν για τα μελλοντικά στάδια και τις διάφορες ε, διαδικασίες και για την ε, τυπολογία των δυνατοτήτων ε, που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την προσέγγιση. Όσον αφορά τις δυνατότητες ε, προγραμματισμού, εμείς είμαστε υπέρ αυτής της επιλογής και θα ήθελα να ξέρω αν αυτή η αξιολόγηση κόστους ωφελίας έχει ξεκινήσει, ε, σκοπεύετε να ξεκινήσετε τη μελέτη τι γίνεται με το χρονοδιάγραμμα και τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτά. Όσον αφορά τώρα τη Λιβύη, θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες για τη διαδικασία ε, δημιουργία συσσόρευσης δυνάμεων για την αποστολή στη Λιβύη και θα συμφωνήσω λίγο και με τους προλαλήσαντες. Υπάρχει μια γενικότερη απογοήτευση και ανησυχία από τη μια ξεκίνησε αποστολή και από την άλλη είναι πολύ περιορισμένη η εντολή της ε, και ίσως ε, δίνουν έναν ακατάλληλο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το θέατρο επιχειρήσεων. Υπό αυτή την έννοια, αν και το θέμα δεν είναι αυστηρά ευρωπαϊκό, αλλά εσείς είστε υπουργό μιας εκ των χωρών που συμμετέχει στην αποστολή του ΝΑΤΟ, θα ήθελα λοιπόν μια σύνθεση για την κατάσταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο κύριος Κυριλόφ, τελευταία ερώτηση, γιατί μετά μόνο 8 λεπτά θα έχουμε για να μας απαντήσει ο υπουργό, οπότε σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, χτες ρώτησα την Επιτρόπο Γεργέωβα για την κακή αυτή κατάσταση όσον αφορά τον κόσμο που βρίσκεται στα βουνά δυτικά της Τρίπολης. Είναι τραγική κατάσταση, τους κάνουν έκκληση για βοήθεια. Ρωτάω λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε με κάποια ανακούφιση εξαίρως ή κάπως αλλιώς, τι προτείνετε. Αυτό τη ρώτησα και είπε ότι θα φτάσει η βοήθεια στα χέρια του Καντάφη τελικά. Εγώ όμως δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Θα βοηθούσε λίγο τον κόσμο που αγωνίζεται κατά του Καντάφη. Δεύτερον, Πόλεμος κατά της πειρατείας. Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά πώς είναι δυνατόν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να μην μπορούμε να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Έχοντας υπόψη μας ότι υπάρχουν ε, και ρωσικά και κινέζικα πλοία. Εδώ τίθεται υποφεσβήτηση η επιτυχία ολόκληρου του εγχειρήματο. Μήπως υπάρχει ένας άλλος τρόπος με διαφορετική ή κάτι άλλο για να έχουμε μια αποτελεσματική δράση. Οι Αμερικανοί μήπως θα μπορούσαν να βοηθήσουν περισσότερο. Κάποιες ε, χώρες λένε ότι ίσως θα έπρεπε να το ξαναδούμε. Μήπως να υπάρχει και κάποια παρέκκληση. Τη στιγμή που έχουμε και την Κίνα και τη Ρωσία θα μπορούσαμε κάτι να αλλάξουμε. Ο Υπουργό, σε 7 λεπτά μπορείτε να απαντήσετε. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομο ε, και από το Συμβούλιο ακόμα. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τόσα είπατε και θα τα μεταφέρω στην κυρία Άστον. Θα απαντήσω συγκεντρωμένα στις ερωτήσεις σας και θα κάνω και κάποιες προτάσεις. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ. Δεύτερον, υπογραμμίζω ότι όπως και εσείς έτσι και εγώ είμαι πάρα πολύ φιλόδοξος για το PST και για την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ. Όπως γνωρίζετε, στα τέλη της Προεδρίας μας σας ενημέρωσα κυρίως για το πλαίσιο της ε, Γάνδης, το περίφημο pooling and sharing, δηλαδή πώς θα μοιραζόμαστε τους πόρους μας, πώς θα τους βάλουμε από κοινού είναι πολύ σημαντικό. Αλλά τίθεται θέμα βούλησης εδώ. Και ίσω το δημοσιονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε να αποτελεί ένα άλοθη τελικά για να μην προχωράμε περισσότερο. Ακούω τα σχόλιά σας για το UTM. Όπως σας είπα θα μεταφέρω τα σχόλιά σας στην είπατε εκπρόσωπο. Άλλος υπουργό Βελγίου σας λέω ότι προσπαθούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με το σύστημα κατάρτισης σε ένα αναγνωρισμένο σύστημα. Μερικές φορές έχουμε παραδείγματα που αναφέρατε κι εσείς. Η συζήτηση τώρα για το UTM στην Σομαλία ξεκίνησε με συζήτηση μεταξύ πρέσβεων. Αύριο θα αποφασίσουμε για το τι συνέχεια θα δώσει το Συμβούλιο. Πρέπει να έχουμε ένα νέο πλαίσιο χωρών γιατί η Ισπανία, για παράδειγμα, αποφάσισε να αποσυρθεί. Για τη Λιβύη. Συμφωνώ με τις παρεμβάσεις που άκουσα. Επιμένω για να επενθυμίσω ότι το Βέλγιο ήταν από τις πρώτες χώρες που συμμετείχε στη συμμαχία με 6 F-16 από την Άραξο στην Ελλάδα και με ένα διοκτικό καταδιοκτικό. Μάλιστα χτες είχα την ευκαιρία να πάω κι εγώ αυτοπροσώπως. Τα μηνύματα τα οποία ακούσαμε εδώ για τη Λιβύη είναι σημαντικά. Όμως ακούστε για το λειτουργικό μήμα Υπάρχει μια ομάδα ειδικών τώρα στην Βεγγάζη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Γκόμες, για να αξιολογήσει τις μελλοντικέ ανάγκες στον τομέα της ασφάλειας και τι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται. Φυσικά και χρειάζεται, οπωσδήποτε, δεδομένων των εμπειριών που μας μεταφέρατε πριν από λίγο. Για την UFOR τώρα. Η εντολή είναι ξεκάθαρη νομίζω. Μπορούμε να δράσουμε μόνο εφόσον το ζητήσουν τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. ευκαιρίες για pooling and sharing φυσικά είναι πολύ σημαντικές και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή που έχουμε τώρα και φιλοδοξίες υπάρχουν. Και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε στην ίδια φιλοδοξία. Έχουμε 300 προγράμματα που έχουν υποβληθεί παραπάνω, μάλιστα. Προτάσεις δηλαδή για pooling and sharing. Θα εξεταστούν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, από την EDA. Εξετάζονται καθημερινά. Τέλη, μάλλον μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουμε ολοκληρώσει τη δουλειά μας εκεί. Τώρα για τον πάρκο όπλων στη Λιβύη ισχύει. Αυτό που ακούω πολύ συχνά και εγώ και οι συνάδελφοι, και εδώ δεν μιλάω μόνο ως πρόσωπος της κυρίας Άστον, αλλά και από τους συναδέρφους. Η αναλογία των μέσων που πηγαίνει στην Αταλάντα σε σχέση με τη σύλληψη πειρατών που πάνε σε δίκη. Υπάρχει ένα νέο σχέδιο δράσεων που θα εγκριθεί με πιο ισχυρές δράσεις και θα συμπεριλάβουμε και την δυνατότητα κινητοποίησης και άλλων ε, σκαφών ε, αντίστοιχων με αυτά που χρησιμοποιούν οι πειρατές. Φυσικά η πρόληψη είναι ό,τι καλύτερο. Και πάνω σε αυτό πρέπει κυρίως να δουλέψουμε. Ξέρουμε ότι η πρόληψη ξεκινάει στην Αφρικανική Ήπειρο. Όλες οι δράσεις χρειάζονται τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Εμείς προστατεύουμε τα πλοία μας επιτυχώς σχετικά και σας μεταφέρω την πεποίθηση της είπα της εκπροσώπου και τη δικιά μου ότι ξέρουμε ότι δεν φτάνει. Δεν είχα περισσότερο χρόνο. Αυτά, Πρόεδρε. Πάντως να ξέρετε ότι λαμβάνω υπόψη μου τις δικές σας συστάσεις. Και ελπίζω ότι θα επανέλθουμε σε μια άλλη συνάντηση. Αλλά τότε να μην ξεκινήσουμε στις 11.30. Ας ξεκινήσουμε στις 10 καλύτερα για να έχουμε περισσότερο χρόνο. Δεν μου απαντήσατε για την φιλοδοξία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Η φιλοδοξία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ε, και του υπευθύνου ήταν σαφής. Είμαστε υπέρ της εργασίας του EDA στο pooling and sharing και αυτό συνάδει με αυτά που φασίστηκαν στη Γάνδη ε, στο άτυπο Συμβούλιο Κορυφής και επιβεβαιώθηκε στο επίσημο Συμβούλιο Κορυφής πέρυσι το Δεκέμβριο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Αμήνης. Και βεβαίως στηρίζουμε ε, την no-fly zone, την ζώνη που δεν επιτρέπεται να γίνεται πτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Και πάλι, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που είχαμε τόσο λίγο χρόνο, ήμασταν πιεσμένοι. Η επόμενη συνεδρίαση θα είναι στις 14 Ιουνίου με μία κρόαση ε, για ε, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσεως ή στα θέματα αμήνης. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και πάλι και ελπίζω να σας ξαναδούμε σύντομα.